Uh, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και τρεις συνάδελφοι που είναι εδώ, θα ξεκινήσει, επαναλαμβάνει τη συνεδρίαση. Έχουμε ανακοινώσεις ε, του Πρόεδρου, γιατί ξεκινήσαμε τρεις και δέκα. Λοιπόν, να σας πω τι έγινε στους συντονιστές. Ε, συναντηθήκαμε να συζητήσουμε τις προτεραιότητες μας για το νομοθετικό πρόγραμμα της Κομισιόν για το 2011. Η απόφασή μας είναι η εξής. Ως συνέχεια του λεγόμενου διαλόγου με τον Αντιπρόεδρο Κάλλας, οι πολιτικές ομάδες εξέθεσαν τις προτεραιότητες τους και αποφάσισαν να υποβάλουν έξι προτεραιότητες ε, εξ ονόματος της Επιτροπής. Αυτές θα είναι αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, μεταξύ των οποίων εφαρμογή, χρηματοδότηση και συνοχή, εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους για όλα τα μέσα μεταφορών για να μειωθεί το διοξίδιο του άνθρακα, ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ εργαζομένων και εταιριών που μπορεί να σημαίνει κοινωνική νομοθεσία οδηγίες ασφάλειας ε, από ατυχήματα και κακόβουλες ε, ενέργειες καθώς και ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και τα δικαιώματα των επιβατών που αλλάζουν μέσα ε, μεταφοράς και ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ε, τουρισμού. Αυτές ήταν οι έξι προτεραιότητες που ομόφωνα ενέκριναν οι συντονιστές σήμερα. Τώρα θα αποστέλουμε μία επιστολή στον πρόεδρο της διάσκεψης ε, των πρόεδρων των επιτροπών και μετά θα εγκριθεί από την διάσκεψη των πρόεδρων ως συνεισφορά του Κοινοβουλίου για το νομοθετικό έργο της Κομισιόν του 2011. Όλοι ικανοποιημένοι, βεβαίω κοιτάω τα έδρανα, όλοι ικανοποιημένοι, είναι ωραία. Στα διάφορα συμφωνήσαμε επίσης πως ο Πρόεδρος θα αποστείλει μια επιστολή στην Κομισιόν ζητώντας να εξεταστεί η επιβολή της κείμενης νομοθεσίας ασφαλείας όσον αφορά τα γεωργικά οχήματα μετά το πρόσφατο ατύχημα στο Βέλγιο που έχασαν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι με, σε ένα ατύχημα μεταξύ ενός γεωργικού ελκυστήρα και ποδηλατών. Ήταν έτοιμα των πρασίνων αυτό και οι συντονιστές ε, συμφώνησαν ο πρόεδρος να αποστείλει την ε, επιστολή αυτή για την επιβολή της κείμενης νομοθεσίας. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις του Προέδρου. Αν είστε όλοι ευχαριστημένοι, περνάμε στο επόμενο σημείο. Δεν ορίσαμε εισηγητές ε, Οπότε περνάμε στην παρουσίαση των προτάσεων της Επιτροπής για τον Προπολογισμό. Και ο εισηγητής είναι ο Αντιπρόεδρος Ενρίκε. Οπότε έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή και κυρίως την Επιτροπή Προϋπολογισμού αλλά και την Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών για την ενάργεια των εγγράφων που διαβιβάστηκαν και για τις συζητήσεις που κάναμε μετά τη δημοσίευση του σχεδίου Προϋπολογισμού. Για συντομία, θέλω να σας πω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, γενικά σε επίπεδο κοινοβουλίου. Τώρα για τις μεταφορές. Χοντρικά, Υπάρχει μια αύξηση κατά 11% των πιστώσεων δεσμεύσεων με μια μείωση 2% των πιστώσεων πληρωμών. Αλλά αυτή η μείωση των πιστώσεων πληρωμών όταν επανερχόμαστε στις, στις μεταφορές πέρα από τα διοικητικά έξοδα φτάνουμε σε 14% αύξηση των πιστώσεων δεσμεύσεων και στο ίδιο νούμερο 1 δισεκατομμύριο 77 δισεκατομμύρια ε, πιστώσεων πληρωμών γιατί η Κομισιόν έκανε μια προσπάθεια και ίδια περιόρισε τα έξοδά της και διατήρησε το ίδιο επίπεδο πιστώσεων πληρωμών μειώντας κατά 3% τα έξοδα τα διοικητικά για τη λειτουργία της. Τη συγχαίρουμε. Τώρα, το ουσιαστικό για τις μεταφορές, γιατί στις ε, πιστώσεις προμών είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Οι δικαιούχοι είναι κάποιες agencies, ιδίω για την ε, ασφάλεια των αέριων μεταφορών και των συντροφικών μεταφορών, μικρή αύξηση. Η υπηρεσία για τις αλλαίσεις μεταφορές είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο, ενώ οι πιστώσεις για την ε, ασφάλεια και τα δικαιώματα των επιβατών μειώθηκαν για να υπάρξει μια προσαρμογή. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα TNT, υπάρχει ουσιαστική αύξηση 180 εκατομμύρια με διατήρηση των πιστώσεων πληρωμών και των αδειών για τις πιστώσεις πληρωμές, ουσιαστική αύξηση για τις πληρωμές στο TNT, διατήρηση του προγράμματος ΣΕΖΑΡ με μικρή αύξηση των πιστώσεων πληρωμών. Ίσως θα υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στο μέλλον και, του, και το Μάρκο Πόλο ε, για τις πιστώσεις πληρωμών έχουμε μικρή μείωση και αύξηση των ε, εγκρίσεων των προγραμμάτων. Προγραμμάτων που μέχρι στιγμής κινήθηκαν καλά, λειτουργήσαν καλά. Αυτά για τις μεταφορές. Χοντρικά υπάρχει μικρή αύξηση για τις α, ε, υπηρεσίες, τα agency, ουσιαστική αύξηση του TNT για την έγκριση των προγραμμάτων και μικρή μείωση για τα υπόλοιπα. Κατά τα λοιπά, ο προπολογισμό είναι πανομοιότυπο. Πανομοιότυπο ε, προπολογισμό της ε, πιστώση ε, πληρωμών σημαίνει συμπίεση ουσιαστικά. Ε, Προπολογισμό λοιπόν λιτότητα, μια μικρή προσπάθεια για τις agencies και μεγαλύτερη προσπάθεια για τα TNT. Υπάρχει πρόβλημα πόρων, το λέμε και το ξαναλέμε από τους, για τους υπολογισμούς που κάναμε για, τους, για τον προπολογισμό 2012-2013 και τις εκτιμήσεις. Υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει κίνδυνος να μειωθούν τα έξοδα για τις agencies ενώ τους έχουμε δώσει από την άλλη νέα καθήκοντα και νέες αρμοδιότητες και είναι, θα είναι δύσκολο να κάνουμε την ίδια προσπάθεια ε, το 2012-2013 για τις εγκρίσεις ε, πληρωμών και τις πιστώσεις πληρωμών. Τώρα, για το πολιετές πρόγραμμα 2007-2013 έχουμε μεγάλη πίεση που από αυτή τη χρονιά θα οδηγήσει σε ε, μια σχετική διατήρηση του προπολογισμού των μεταφορών. Ε, για το 12-13 προοπτικές δεν είναι πολύ καλές και τεράστιες δυσκολίες για να εφαρμόσουμε νέες πολιτικές της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής αυτής μεταφορών. Ε, η μόνη ελπίδα που μπορούμε να έχουμε αφορά μια αύξηση των μέσων. Ε, τρία είδη μέτρων δηλαδή σημαίνει αυτό. Είτε αναθεώρηση του πολιετούς πλαισίου, αλλά ξέρουμε ότι το Συμβούλιο ανθίσταται και υπάρχει διελκυστίνδα με τις ταξίδες της Επιτροπής Προπολογισμού και του Συμβουλίου. Εξάλλου το Συμβούλιο καθυστέρησε κατά ένα χρόνο την αναθεώρηση αυτού του πλαισίου και αν δεν υπάρξει αναθεώρηση του πλαισίου, δεν θα υπάρξει αύξηση των αιτησιών πόρων και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή που θα γίνει φέτο. Έχουμε δύο άλλου τρόπου για να αυξήσουμε τα μέσα μα. Ο πρώτο είναι να ενεργοποιήσουμε διαφορετικά τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά ταμεία. Για τα περιφερειακά ταμεία να ζητήσουμε να υπάρξει προτίμηση και να δοθούν κονδύλια κυρίω στι υποδομέ που συνδέονται με τα TNT από το να αφήσουμε τα κράτη να προωθήσουν ε, οι υποδομές που δεν έχουν ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, να τα κινητοποιήσουμε για να στραφούν προς ε, ε, προγράμματα ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Και τρίτος τρόπος είναι νέα μέσα, είτε ειδικό ταμείο για τις μεταφορές, αναφέρθηκε αυτή η ιδέα εδώ, είτε να έχουμε άλλα έσοδα για υποδομές ευρωπαϊκού χαρακτήρα, είτε χρησιμοποιώντας οικονομικά και χρηματοδοτικά μέσα, αλλά η, χρηματοδο... η χρήση τέτοιων ειδικών πόρων όπως τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες Επενδύσεων δεν είναι προσπελάσιμα από το Κοινοβούλιο γιατί δεν έχουμε ιδίους πόρους και επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο άμεσα. Επομένως, ε, πρόβλημα με τον προϋπολογισμό ε, έκανε όμως την προσπάθειά της η Κομισιόν έκανε θυσίε σε ό,τι αφορά τα διοικητικά έξοδα, αλλά το μέλλον είναι αβέβαιο. Για τον προπολογισμό τουρισμού. Δεν συμμετείχα, δεν θέλησα να συμμετάσχω στις συζητήσει για τον τουρισμό και τα συναφή θέματα, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει πρόβλημα με τον προπολογισμό τουρισμού. Γιατί δεν υπάρχει βασικά ένα τέτοιο προπολογισμό. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν. Μπορείτε να βρείτε δημοσιονομικές γραμμές για τον τουρισμό μόνο εκτός, από αυτής της Επιτροπής που ουσιαστικά έχει την ευθύνη. Οι ελάχιστες γραμμές προπολογισμού που μπορούν να πάνε για τον τουρισμό, για τον τουρισμό βρίσκονται στην, στα χέρια της Επιτροπής Ήτρε και στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση στα πλαίσια ενός υποπρογράμματος 6 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα ΕΑΗ, αλλά δεν είναι δική μας αυτή η δημοσιονομική γραμμή. Έχουμε την αρμοδιότητα, αλλά χρήματα λοιπόν. Ο μόνος τρόπος να παρέμβουμε στα, στο πρόβλημα αυτό του προπολογισμού του τουρισμού είναι μέσω πιλωτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων δράσης. Αναφέρθηκαν κατά επανάληψη σήμερα το πρωί, πράγματος χάρη το καλυψώ. Αλλά τα τρία προγράμματα που έχουμε τελειώνουν το 2011. Έχουμε δύο πιλωτικά πρόγραμματα ε, για τις μεταφορές, δεν θα μιλήσω για αυτά, ενώ για τον τουρισμό δεν έχουμε τέτοια πιλωτικά προγράμματα. Επομένως, ζητώ από τα πολυάριθμα μέλη της Επιτροπής που είναι παρόντα σήμερα να συνεισφέρουν α, σύντομα, γιατί οι προθεσμίες είναι σφιχτές, ε, για τα πιλωτικά προγράμματα και, τα, και τις πιλωτικές δράσεις ε, και τα σχέδια δράσης. Πολύ σύντομα λοιπόν πρόεδρε, άμα επιτρέπετε τώρα να σας δώσω μια ιδέα για την ατζέντα μας, που και αυτή είναι πιεστική. Η Επιτροπή και ο προπολογισμό έγιναν καθυστερημένα. Στα πλαίσια επίσης της Λισαβόνας έχουμε μόνο μια ανάγνωση. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόγραμμα, να σας αναφέρω η Επιτροπή, ο εισηγητή προπολογισμού, τμήμα 3, στην Επιτροπή Προπολογισμού θα παρουσιάσει μία έκθεση στις 5 Μαΐου. Καταρχήν θα, θα υποβάλει την έκθεση στις 5 Μαΐου και θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Προπολογισμού στις 10 Μαΐου και η καταληκτική ημερομηνία για τις οπολογίες θα είναι η 12 Μαΐου. Το λέω στους σκιώδεις ε, εισηγητές. Ε, μεταξύ 10 και 12 Μαΐου εκεί πρέπει να κινηθούμε. Έχουμε 48 ώρες. Αυτή η έκθεση θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμού στις 2 Ιουνίου και υπενθυμίζω ότι η κοινοβουλευτική ψηφοφορία για το ψήφισμα θα γίνει στις 15 Ιουνίου. Βλέπετε ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ πιεστικό για αυτό το ψήφισμα της Επιτροπής Προπολογισμού. Ε, και εμεί θα πρέπει να συνεισφέρουμε παρόλα αυτά σε αυτό. Έχουμε τη 15η Ιουνίου τη θέση του, του Συμβουλίου για την πρόταση προπολογισμού τη Επιτροπής στι 8 Σεπτεμβρίου για τι επιτροπέ, δηλαδή για εμά και τα μέλη, του βουλευτέ, 13 ε, Σεπτεμβρίου τις, ε, στις πολιτικές Αυτέ ομάδες. Αυτές είναι οι καταρτικέ ημερομηνίες για τις τροπολογίες. 30 Σεπτεμβρίου ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμού και στις 18 με 22 ψηφίζει το Κοινοβούλιο. Συνοψίζω. Για τις τροπολογίες στο σχέδιο ψηφίσματος μεταξύ 10 και 12 Μαΐου έχει δυνατότητα να παρέμβετε. Επίσης, ε, μέσα αυτή την, ε, σε αυτό το διάστημα θα γίνουν προτάσεις, θα πρέπει να γίνουν προτάσεις για τα πιλωτικά προγράμματα και τα σχέδια δράσης. Η θέση του Συμβουλίου θα την ξέρουμε στις 15 Ιουνίου, τότε που φεύγουν όλοι οι διακοπές. Μην ξεχνάτε ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να, γίνουν, να έχουν κρατηθεί το αρχότερο μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου. Έτσι. Ε, μην ξεχνάτε τις ημερομηνίε, είναι σημαντικές. Ε, θα είναι δύσκολο να δουλέψουμε δεδομένου του πιεστικού χρονοδιαγράμματος. Είναι σημαντικό όμως να συνεισφέρουμε, γιατί στο πρώτο ψήφισμα της Επιτροπής Προπολογισμού, χάρη στη δουλειά που έγινε από τα μέλη της Επιτροπής, ακουστήκαμε, Αλλιώ θα είχαν εξαφανιστεί οι μεταφορές, επομένως ε, προσέξτε την, ε, το τελικό ψήφισμα τη Επιτροπή Προπολογισμών για τον ίδιο λόγο γιατί είμαστε σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο πολύ λιτό, πολύ πιεστικό. Ζητώ λοιπόν από τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και από τους σκιώδεις συζητητές να σκεφτούν τις προοπτικές του 2012-2013. Έχουμε πίεση χρόνου, έτσι, το λέω για τις τροπολογίες και τεράστιες δημοσιονομικές πιέσεις. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Μπενούτσι από την Κομισιόν. Θα θέλατε να μας παρουσιάσετε την άποψη της Κομισιόν για αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον αντιπρόσωπο, τον αντιπρόεδρο, συγγνώμη, και εισηγητή. Στα γαλλικά συνεχίζω. Νομίζω ότι ο συγγητής συνόψε σωστά την κατάσταση Πρέπει να κάνουμε λοιπόν κάποια πειθαρχία και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε ο προπολογισμό του 2011 να μην ξεπεράσει το πλαφόν που προτείνει ο μακροχρόνιος προγραμματισμός μέχρι το 2013. Και εσείς διαπιστώσατε μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προγράμματα Trans-European Network που χρειάζονται γύρω στο 14% που αυξάνονται νομίζω κατά 14%. Έχουμε κάποιες μικρές μετακινήσεις για τις υπόλοιπε γραμμές. Για το πρόγραμμα λέω, η Γενική Διεύθυνση έχασε την διεύθυνσή του και το GOC που πέρασε στην διεύθυνση για τις επιχειρήσεις. Όσον, όσον αφορά τη μικρή διαφορά που διαπιστώσατε εσείς μεταξύ πιστώσεων δεσμεύσεων και πιστώσεων πληρωμών θα έπρεπε να διευκρινίσω ότι οι πιστώσεις πληρωμών αντανακλούν την ταχύτητα εφαρμογής του προγράμματος. Η Κομισιόν λοιπόν πληρώνει όταν φτάνει το τιμολόγιο. Αντίθετα, οι πιστώσεις δεσμεύσεων αποτελούν ένα έδος υπόσχεσης και δυνατότητας η Κομισιόν για το επόμενο υψηλότερο πλαφόν όταν θα συναυθεί η σύμβαση. Να επανέλθω γρήγορα στα υπόλοιπα προγράμματα. Μάρκο Πόλο, Σεζάρ, που έχουν διατηρηθεί περίπου. Το Μάρκο Πόλο λειτουργεί καλά. Οπότε συνεχίζουμε να το τροφοδοτούμε και ελπίζουμε η χρηματοοικονομική κρίση να μην έχει επιπτώσεις στην εφαρμογή αυτής της δουλειάς που έγινε το 2008 και 2009. Για το ΣΕΖΑΡ διατηρήσαμε το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης. Η κατάσταση λοιπόν είναι περίπου αμετάβλητη. Και υπάρχει ένα στοιχείο για το οποίο θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σας. Η δυσκολία που συνάντησε η Γενική Διεύθυνση για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των υπηρεσιών δεν είναι πρώτη φορά. Ξέρουμε ότι αυτές οι υπηρεσίες από το 2007 έχουν αναλάβει την υποστήριξη της εφαρμογής των προγραμμάτων και το έργο ικανοποίηση των ετοιμάτων αρρωγής της Μητρικής Γενικής Διεύθυνσης και αυτό επιφέρει ένα σημαντικό οικονομικό φόρτο. Ικανοποίησαμε λοιπόν αυτά τα αιτήματα έχοντας δύο μοχλούς. Καταρχήν την κατανόηση των αιτημάτων τους και δεύτερον προσπάθεια ικανοποίησης τους με αντιστάθμιση δικαιολογημένων δαπανών όπου υπήρχε νομική βάση και όπου εγκρίθηκε δηλαδή από το Κοινοβούλιο αναζητώντας ε, τις πιστώσεις από άλλες γραμμές. Δηλαδή στα γαλλικά όπως τα λέγαμε αποψηλώσαμε τις ε, γραμμές που ήταν γραμμές υποστήριξης σε άλλα σημεία και έστω και αν δεν ικανοποίησαμε πλήρως τα αιτήματα όλων των υπηρεσιών. Η υπηρεσία, ας πούμε, για τους ιδεοδρόμους αλεάζα κλπ. κλπ. Για το 2012 λοιπόν και 2013 θα πρέπει να εξετάσουμε εδώ, σε αυτή την Επιτροπή δηλαδή, το κατά πόσο θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να αποψηλώνουμε αυτές τις γραμμές που συνεχίζουν να φτάνουν σε μια κριτική μάσα ή αντίθετα να βρούμε άλλες πηγές χρηματοδότησης ακολουθώντας τάξεις μεγέθους από 20 εκατομμύρια ευρώ για να φτάσουμε σε αυτές τις χρηματοοικονομικές ε, προοπτικές ώστε να καλύψουμε τα αιτήματα των υπηρεσιών για τις οποίες έχουμε αρμοδιότητα. Εκεί λοιπόν σημαίνει ότι θα μπορέσουμε πια να απευθυνθούμε σε γραμμές όπως οδική ασφάλεια ή σε γραμμές υποστήριξης στις οποίες είχαμε βασιστεί μέχρι τώρα. Θα πρέπει δηλαδή να βρούμε κάποια άλλα στοιχεία Ο κ. Ε, Καλοφελίπε προτείνει δεχομένω να χρησιμοποιήσουμε το περιθώριο ή να βρούμε άλλους τρόπους. Αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε και θα πρέπει ενδεχομένω να κάνουμε και μια αξιολόγηση των πιο ενδιαφερόντων προγραμμάτων προγράμματα που ενδεχομένως φτάνουν στην ορίμανσή τους. Ίσως εκεί λοιπόν θα μπορούσαμε να οικονομήσουμε, εξοικονομήσουμε, να πάρουμε κάποιο μικρό ποσό και να καλύψουμε τις ανάγκες μας αλλού για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι φυσιολογικό να εφιστήσω δηλαδή την προσοχή σας ε, σε αυτό το θέμα που αφορά και χαρακτηρίζει νομίζω το προγραμματισμό για το 2011. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λιμπεράτσικη. Mr. Chairman ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας δώσατε μία σαφή εικόνα της κατάστασης την οποία επιβεβαίωσε και ο κύριος Μπονούτσι. Πραγματικά η κατάσταση έχει όπως έχει. Οι απόψεις μου βεβαίως είναι προσωπικές αυτή την στιγμή και όχι ίσως ομάδας μου. Το μέλλον του προϋπολογισμού είναι όλο και λιγότερη ευελιξία. Έχουμε τα άκαμπτα έξοδα. Οπότε το ερώτημα είναι ποιος είναι ο ρόλος του προϋπολογισμού. Απλά θα χρηματοδοτούμε την καθημερινή λειτουργία ή θα έχουμε ξανά έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα χρηματοδοτεί νέα προγράμματα και πρωτοβουλίες δεν είναι τόσο προφανές το δεύτερο. Φοβάμαι πως είναι πολύ περιορισμένο και είναι θεμελιώδες αυτό το ερώτημα. Ίσως, κύριε Πρόεδρε, καμιά φορά θα έπρεπε να καθίσουμε να πιούμε έναν καφέ και να συζητήσουμε ποιο θα είναι το μέλλον, ειδικά το 2012-2013. Η επιλογή που ανέφερε ο κύριος Ρικέ. Θυμάμαι που ε, στο παρελθόν μιλούσαμε για διαρθρωτικά ε, ταμεία και ταμεία συνοχής και το κομμάτι των μεταφορών. Απ' τη μία παρατηρούμε πως τα διαρθρωτικά τα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών έχουν αυξηθεί κατά 14% αλλά υπενθυμίζω πως είναι μόνο 180 εκατομμύρια να σας υπενθυμίσω πως εμείς ε, αναμέναμε 23 δισεκατομμύρια και πήραμε 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάπως λιγότερα από όσα περιμέναμε. Θα γίνει λοιπόν μια ενδιάμεση αναθεώρηση των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων συνοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες 18 Μαρτίου, τρέχοντος τους Γύρω στο 16% των συνολικών κονδυλίων συνεχής είναι ήδη ε, έχουν είναι ήδη στην κατηγορία των πληρωμών, χωρίς να σημαίνει αυτό πως έχουν χρησιμοποιηθεί. Ο χρόνος περνάει, οπότε ήδη έχει περάσει ο μισός χρόνος των προοπτικών 2007-2013 και έχουμε εξοδέψει ένα 16% μόνο των ποσών. Οπότε ίσως έχετε δίκιο. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα θέματα. Δηλαδή ικανότητα απορρόφησης. Να δούμε που έχουμε κάποια πιθανότητα και ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας για το πώς περιμένουμε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια. Επίσης, συμφωνώ πως θα πρέπει ίσως να μιλήσουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Αυτά είναι τα σχόλιά μου για να βρούμε μια διέξοδο. Για να επανέλθω τώρα στο θέμα. Πράγματι δεν είναι το θέμα οι μήνες και τα έτη. Πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική αλλαγή στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για τους σιδηρόδρομους, για τις αερομεταφορές, τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Το να κρατήσουμε το Μάρκο Πόλο και να δούμε κάποιες δυνατότητες ξεκονόμησης π.χ. το 3% των λειτουργικών δαπανών της ε, Κομισιόν είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά Νομίζω πως θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα πιλωτικά αυτά προγράμματα. Θα μπορούσαμε ίσως να λάβουμε κάποια πράγματα υπόψη για εμάς. Είναι προτεραιότητα οι μεταφορές και η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη. And ε, πώς θα αντιδράσουμε. Και ε, ειλικρινά δεν έχω τίποτα να προσθέσω αυτή τη στιγμή. Γιατί καλά τα πήγε ο εισηγητής. θα έπρεπε να έχουμε νομίζω περισσότερο χρόνο να το συζητήσουμε εισηγητής και σκιώδης αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Ευχαριστώ η κυρία Γένσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Ρικέ που μας είπε πόσο δύσκολα προδιαγράφονται τα πράγματα για τον προπολογισμό. Είναι λυπηρή κατάσταση καθώς έχει πολύ αυστηρά όρια, έχουν πολύ αυστηρά όρια μεταφορές και φαίνεται πως ε, το 2011 το περιθώριο θα χρησιμοποιηθεί για τις νέες ε, αποκεντρωμένες υπηρεσίες στον, δημοσιο... στον χρηματοοικονομικό τομέα. Και τα επόμενα χρόνια μας λέει ήδη η Κομισιόν πως είναι αρνητικό το περιθώριο λόγω των έργων αυτών των ε, ETR. Οπότε είναι δύσκολη η κατάσταση και συγκεκριμένα νομίζω είναι λυπηρό πως οι υπηρεσίες έχουν βρεθεί στην κατάσταση που μας περιέγραψε η Κομισιόν. Οι υπηρεσίες αυτές ε, παίζουν ε, σημαντικό ρόλο για την πολιτική μεταφορών ε, και στην ασφάλεια και είναι κρίμα να έχουν αυτούς τους αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς ρωτήσαμε από πού θα μπορούσαν να βρεθούν τα χρήματα και πώς θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα. Χρειάζεται νομίζω αυτή η μεσοπρόθεσμη θεώρηση και να εξετάσουμε τα πράγματα. Ο κύριος Λιμπεράτσκι ανέφερε το θέμα των διαρθρωτικών ταμείων. Πολιτικά θα είναι δύσκολο να πάρουμε λεφτά από τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά θα βρεθούμε σε μια κατάσταση της ε, ρήτρας ε, σταδιακής κατάργησης και Εκεί έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια χρήση αυτών των κονδυλίων για άλλους σκοπούς. Αλλά νομίζω πως πρέπει να δούμε και τις δικές μας αρμοδιότητες. Παράδειγμα τους χάρη δεν μπορούσαμε να εξοδέψουμε όλα τα κονδύλια του Μάρκο Πόλο, οι κανονισμοί άλλαξαν. Αλλά είναι ενδιαφέρον νομίζω το ότι δεν μπορούμε να εξοδέψουμε τα χρήματα του Πόλο ενώ Κάθε χρόνο υπάρχουν πάρα πολλά καλά έργα στα διευρωπαϊκά δικτύα μεταφορών και στις αιτήσει από διαθέσιμα κονδύλια. Νομίζω λοιπόν πως ε, τα ε, έργα αυτά, τα αιτήσια, είναι και αυτά πράγματα που θα μπορέσουν να μεταφέρουν, ε, να μετατοπίσουν τις μεταφορές από τον από τους δρόμους στη θάλασσα και το σιδηρόδρομο και σε άλλα λιμάνια, ίσως ενδοχώρας και τέτοια. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λίγα κονδύλια παραπάνω για τα διευρωπαϊκά αυτοδίκτυα μεταφορών. Τώρα για τα πιλωτικά έργα θα είναι δύσκολα τα πράγματα δεδομένων των περιορισμών για οποιοδήποτε πιλωτικό έργο. Συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ρικέ για τον τουρισμό. Μπορούμε έτσι να ξεκινήσουμε κάτι. προσπάθησα εγώ να ξεκινήσω ένα πιλωτικό έργο για τη μεταφορά των ζώων στο κομμάτι των προπολογισμών που είναι στη γεωργία. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα ένα περιθώριο, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Και νομίζω πως είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία η, η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καναλτών δεν έχει συνηθίσει σε τέτοια έργα όπως ε, η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών που είναι πολύ πιο έμπειροι. Και γι' αυτό δεν τσουλάει το πράγμα. Αλλά είναι κάτι που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε, δηλαδή πως η μεταφορά των ζώων ε, είναι κάτι που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε για να δούμε βέλτιστες πρακτικές. Βεβαίω είναι ένα γεωργικό ζήτημα, αλλά είναι και ένα ζήτημα μεταφορών. Και οπωσδήποτε απασχολεί τους ανθρώπους αυτό και πρέπει να κάνουμε κάτι. Να προωθήσουμε δηλαδή και την εφαρμογή της νομοθεσίας και να δούμε βέλτιστες πρακτικές. Τέλος, ένα ερώτημα επί της διαδικασίας, γιατί δεδομένου του ότι το χρονοδιάγραμμα είναι τόσο πιεσμένο, προτείνω να στείλετε κατευθείαν τις τροπολογίες στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Ε, κύριε Δικέ, είστε και εκεί μέλος. Όχι. Εντάξει. Θα δούμε τότε. Ε, θα κάνουμε μια γνωμοδότηση. Ωραία. Οπότε υπάρχει η δυνατότητα να συζητήσετε μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Προπολογισμού. Ωραία. Ευχαριστώ. Κύριε Καντσιάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Δεν νομίζω ότι ικανοποιήθηκα με τη δουλειά που έγινε πέραν του γεγονός ότι πρέπει να χρονοτριβήσουμε, πρέπει να παίξουμε και με πόρους που είναι πραγματικά ελάχιστοι. Ε, τρία σημεία για την χρηματοδότηση των θεμάτων μας, τα που, αφορούν, που αφορούν βεβαίως τα αντιευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Γιατί οι υπηρεσίες, οι agencies, με κάποιο τρόπο τέλο πάντων χρηματοδοτούνται. Η μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι στην πολιτική μεταφορών. Αυτή τη στιγμή ακούγονται σημαντικά επιχειρήματα, αλλά αν δεν αλλάξουμε την πολιτική προϋπολογισμού, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει το πράγμα στο μέλλον και δεν θα δώσουμε τις απαντήσεις που οι, χώρα, οι χώρες και η Ευρώπη περιμένουν. Μιλάω για τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και τα νέα εργαλεία. Υπάρχει το αποθεματικό το Μάργκεριτ, το οποίο ποτέ όμως δεν το λαμβάνεται υπόψη. Παρότι δεν αφορά αποκλειστικά τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, αλλά συμπεριλαμβάνει και την ενέργεια μπορεί να ληφθεί υπόψη για να προωθηθούν τα δικά μας θέματα. Κοιτάξτε, είτε θα δημιουργήσουμε ε, άλλα εργαλεία ή θα δημιουργήσουμε τα μέσα που, συζητήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Πρέπει να το συζητήσουμε διεξοδικά αυτό το θέμα. Το δεύτερο, η δεύτερη συνιστόσα της ε, χρηματοδότησης είναι ότι θα πρέπει να προωθήσουμε όλο και περισσότερο τα προγραμματα εταιρική εταιρικής σχέσης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Είναι εκ των ονουκάνευ, γιατί ε, δεν υπάρχουν ακόμα πολλά ε, δημόσια κονδύλια. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τα κράτη-μέλη να αυξήσουν ε, τη συνεισφορά τους. Δεν υπάρχουν λεφτά. Αποκλείεται να διευτευθούν κονδύλια προς την Ευρώπη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το άλλο θέμα είναι ο τουρισμός. Μετά τη Λισαβόνα, ο τουρισμός έγινε, όπως ακούσαμε σήμερα το πρωί, η τρίτη πιο σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα της Ευρώπης. Εμείς διαχειριζόμαστε αυτό το τομέα μαζί με τις μεταφορές. Αλλά δεν έχουμε την αρμοδιότητα για τον προπολογισμό του, του, του, τουρισμού. Θα πρέπει να, λοιπόν, να ζητήσουμε λιμοσύνη από την Επιτροπή Ήτρε, όπως είπατε, ή από τη Γενική Διεύθυνση, που είναι επίσης καθήλυνα αρμόδια ή μέσω των αρμοδίων προγραμμάτων. Αλλά κοιτάξτε, είναι η τρίτη υποτίθεται οικονομική δραστηριότητα. Κάπω θα πρέπει να τη χρηματοδοτήσουμε, το σκεφτούμε και αυτό. Ευχαριστώ, κύριο Αλχαντράουι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν είμαι ειδικό του προπολογισμού και των αριθμών, δεν έχω εμβαθύνει. Και ξέρω πω ε, πράγματι ο συνάδελφο εδώ πέρα μα πέρα με πράγματα από πλευρά ε, επιτροπή ε, του προπολογισμού, αλλά ω επιτροπή μεταφορών θα πρέπει να φύγουμε λίγο από τον τωρινό προπολογισμό να δούμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για το πώς θα μπορέσουν οι προτεραιότητες μας να μεταφραστούν σε προπολογισμό. Και αυτό είναι πιο σημαντικό γιατί θα ξεκινήσει η συζήτηση για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο από το 2014 και εκεί πέρα θα είναι η στιγμή της αλήθειας. Θα έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τη Λευκή Βίβλο, το μέλλον των μεταφορών. Συμφωνούμε νομίζω στα μεγάλα και στα σημαντικά θα πρέπει να έχουμε αυτή την αποτελεσματική συντροπικότητα όπως την είπε ο συνάδελφος ο κύριος Ματιέ Γκρός. Αυτό βεβαίως έχει κάποιες ε, συνέπειες. Θα πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των τρόπων ε, μεταφοράς και εντός ε, των μέσων μεταφοράς και αυτό σημαίνει επενδύσεις. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε μαζί με την Κομισιόν ποια μέσα διαθέτουμε έτσι ώστε εντό λογικών πλαισίων να γίνει αυτή η αλλαγή στα δίκτυα των μεταφορών. Και βέβαια θα είναι σκληρή διαπραγμάτευση με τους συναδέλφους της Επιτροπής Ευρωπολογισμού και των άλλων επιτροπών, αλλά τουλάχιστον θα ξέρουμε πού βαδίζουμε. Αυτό θα ήθελα εγώ να ζητήσω και αυτό μπορεί να γίνει ίσως υπό την δική σας ηγεσία και την καθοδήγηση του Προέδρου. Γιατί θα είναι ουσιαστικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ναι, πράγματι. Αυτή είναι η δουλειά των ανθρώπων του προπολογισμού. κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ. Όπως και ο κύριος Χαντραουή, έτσι και εγώ δεν είμαι ειδική επί του προϋπολογισμού, αλλά πάντα είναι η αλήθεια η ώρα της αλήθειας ε, ο προϋπολογισμός. Είχαμε πολλά σχέδια στο παρελθόν. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για τις προτεραιότητές μας και το που θέλουμε να πάμε και πάντα λέμε πως πρέπει να βρούμε πηγές χρηματοδότησης για, για να επιτύχουμε αυτά τα οποία θέλουμε. δι χρημάτων. Ο δε κύριος Επίτροπος ανέφερε πως ε, θέλει να συσταθεί ένα ταμείο συγκοινωνιών, κάτι το οποίο βεβαίως ε, δεν είναι κάτι τόσο απλό. Οπότε δεν ξέρω, έχουμε συνεννοηθεί με την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γιατί εμένα όλα αυτά μου ακούγονται ευχολόγια και δεν βλέπω τίποτα στην πραγματικότητα. εντάξει, ωραία να λέμε ότι θέλουμε κονδύλια, αλλά πούντα και πώς. Δηλαδή το ένα είναι αυτό και Δεύτερον, σήμερα το πρωί ήρθε εδώ πέρα ο κύριο Σταγιάννη, μίλησε για τον τουρισμό και εκεί πέρα μίλησε για λεφτά και είπε πως ε, θέλει να φροντίσει να μπορέσουν να συγχωνευτούν διάφορες γραμμές του προπολογισμού για να έχει μια μεγαλύτερη γραμμή να μπορεί να χρηματοδοτεί διάφορα έργα. Για μένα το ερώτημα είναι αν έχουμε την δυνατότητα να δηλώσουμε ένα πιλωτικό έργο για τον τουρισμό, πόσα λεφτά θα είχαμε. Για να δούμε δηλαδή αν είναι λογικό και ε, να δούμε αν υπάρχουν και τα απαιτούμενα κονδύλια και αν είναι πόσα είναι αυτά πριν αρχίσουμε να εξετάζουμε έργα. Αυτό ερώτημα μιας που δεν είναι ειδική στον προϋπολογισμό. Μάλιστα σας ευχαριστώ. Πρέπει να ακούσουμε και τον κύριο Όλτουν από την πλευρά του τουρισμού να πω και εγώ κάποια πράγματα. Ούτε και εγώ είμαι ειδικό, αλλά νομίζω πως είναι η 19η συζήτηση για τον προπολογισμό που ζω στο Κοινοβούλιο. Να σου πω ότι έγινε τις προηγούμενες 18 φορές και θα γίνει και τώρα. Ό,τι προτείνουμε θα περικοπεί ως ένα βαθμό από την Επιτροπή Προπολογισμού. Αυτός είναι ο ρόλος του στη ζωή. Οπότε το μυστικό της επιτυχίας είναι να ζητήσουμε παραπάνω για να μας περικόψουν και να βρεθούμε εκεί που θέλουμε. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Αντιλαμβάνομαι πως αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα βεβαίως. Αλλά δεν ανάγκη να κάνουμε εμεί τη δουλειά της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Να είστε σίγουροι πως η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα περικόψει από εδώ και από εκεί χωρίς να τους δώσουμε και εμείς βοήθεια. Και μπορείτε να ρωτήσετε και τους συναδέλφους που είναι εδώ από την Επιτροπή Προπολισμού, θα το επιβεβαιώσουν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι σαν το επιχείρημα με τους υπουργού Μεταφορών. Οι Υπουργοί Μεταφορών θέλουν να φτιάξουν το χ, πράγμα, να κάνουν το ένα το άλλο. Και μετά τον γίνονται Υπουργοί Οικονομικών, κάποιος τους γυρνάει το κουμπάκι εκεί πέρα και δεν υπάρχουν χρήματα για να κάνουν τα έργα που ήθελαν οι ίδιοι όταν ήταν Υπουργοί Μεταφορών. Οπότε πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Οπότε εγώ λέω να ζητήσουμε παραπάνω. Ό,τι θέλετε ζητήστε. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Πρέπει να δούμε κάποια έργα και να δούμε βεβαίως εάν ε, τα λεφτά μας φτιάνουν τόπο. Και από αυτή την έννοια πρέπει να δούμε και κάποιες από τις ιερές μας αγελάδες. Και να δούμε ποιά είναι τα λεφτά μας τόπο. Π.χ. ο Μάρκο Πόλο μου έρχεται εδώ πέρα στο μυαλό. Λεφτά δίνουμε αλλά ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πώς προχωράνε οι στόχοι αυτού του προγράμματος. Οπότε νομίζω πως υπάρχει εδώ πέρα ένα πεδίο να δούμε αν πιάνουν τα λεφτά μας τόπο αλλά πρέπει και να είμαστε έτσι πιο ριζοσπαστικοί και εριστικοί αν θέλετε, να ζητήσουμε λεφτά. Ειδικά στον τομέα του τουρισμού που έχουμε τώρα μια νομική βάση. Κάθε φορά που ζητούσαμε λεφτά για τον τουρισμό στο παρελθόν, ο Γιαρζεμπόφσκι εκεί πέρα το έβλεπε γιατί δεν του αρέσει ο τουρισμός. Και το έκοβαν και στην Επιτροπή Προπολογισμού γιατί δεν υπήρχε νομική βάση για τον τουρισμό. Οπότε εύκολα κόβεται. Και κατανοητό. Τώρα υπάρχει νομική βάση, πρέπει να μπει κάτι για τον τουρισμό. Α, και ας το σβήσουν. Ακόμα και αν τους δώσουμε κάτι να κόψουν, εμείς κάνουμε την δήλωση εκ μέρου του τουρισμού και προτείνω να κάνουμε ένα πιλωτικό έργο για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τουρισμό. Μπορούμε να πάμε λίγο παραπέρα και σε αυτό που μου αρέσει εμένα. Πιλωτικό έργο για τις βέλτιστες πρακτικές στην εκπαίδευση ιστορικών μεταφορών. Για να πάει η Κομισιόν προς τα εκεί που τις λέμε, στη βιομηχανική κληρονομιά. Και ας είναι μόνο 100.000 ευρώ. Ας μπει αυτό στον προπολογισμό Ντομινίκ, και να δούμε τι θα κάνουν. Πιλωτικό έργο στον τουρισμό για τη βέλστη πρακτική εκπαίδευση στην ε, κληρονομιά των μεταφορών. Από το περάσουμε όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά τουλάχιστον λέμε εδώ πέρα εκ μέρους του τουρισμού ότι δεν μπορεί να μείνει στην απέξω. Και αυτή τη φορά δεν μπορούν να γυρίσουν να μας πούνε δεν υπάρχει νομική βάση. Γιατί τώρα με, τη βάση, με την συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε κάποια νομική βάση. Οπότε ας το δοκιμάσουμε αυτό, Ντομινίκ. Να δούμε εκεί ποιο είναι το κλίμα. Αλλά να είστε τολμηροί, ζητήστε. Και ούκαν λάβετε βεβαίως. Αλλά εάν το ρίξετε, αν ρίξετε εσείς ήδη τα ποσά, θα τα κόψει ακόμη περισσότερο η Επιτροπή Προπολογισμού και μετά έρχεται και το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θέλει να κάνει τα πάντα χωρίς λεφτά. Το γνωρίζουμε αυτό με την ασφάλεια. Μόλις αναφέρουμε τη λέξη κόστος, παθαίνουν όλοι καρδιακή προσβολή και πέφτουν ανάσκελα. Οπότε ας πούμε, εμείς αυτό θεωρούμε ότι είναι η κατάλληλη πορεία για τις ευρωπαϊκές μεταφορές και τον τουρισμό και καμιά φορά πρέπει εκτός από τα λόγια να έχουμε και έργα, δηλαδή λεφτά. Αυτή είναι λοιπόν η δική μου η συμβουλή, επειδή δεν είμαι ειδικό στον προπολογισμό, αλλά έχω 19 χρόνια εμπειρίας του προπολογισμού εδώ μέσα. Κύριε θέλετε να μας πείτε και σε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να διευκρινίσω κάποια πράγματα σχέση με το 2011. Το προσχέδιο προπολογισμού που ξεκινήσαμε να συζητάμε σήμερα να σας ενημερώσω επειδή δεν φαίνεται ξεκάθαρα από το προσχέδιο της Κομισιόν για τον τουρισμό. Όπως ξέρετε για το 2010 είχαμε δύο είδη δράσεων. Ένα είδος που χρηματοδοτούσαμε μέσω του προγράμματος επιχείρηση και κοινοτομία και πέρσι, μάλλον και φέτος, θα δώσουμε γύρω στο 1 εκατομμύριο και είχαμε και τις τρεις προπαρασκευαστικές δράσεις που είχαμε προωθήσει πριν από λίγα χρόνια, τρία-τέσσερα περίπου, για τους φορακούς προορισμούς ε, αριστείας και τα άλλα δύο κοινωνικός τουρισμός, καλύψω και διαδρομές ποδηλατοτουρισμού ισχύουν για το 11 υπό τον όρο βέβαια ότι η Κομισιόν δεν αλλάζει τα ποσά για το PM και τις δράσεις του για τον επόμενο έτος μαζί με τα ποσά που θα δώσουμε του χρόνου για, αυτά, για αυτούς τους τομείς στον τουρισμό θα αυξήσουμε και τα κονδύλια από 1 σε 6 εκατομμύρια και όπως είπε ο κύριος Σταγιάννη αυτό θα γίνει στα πλαίσια του προγράμματος της καινοτομία και την επιχειρηματικότητα για το 2011. Αυτό για να περιλάβουμε τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του ΙΔΕΝ, της ΕΔΕΜ δηλαδή, του προγράμματος ΕΔΕΜ και σε σχέση με την ανακοίνωση της Κομισιόν που θα βγει τον Ιούνιο. Αυτά για το 2011. Βεβαίως θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες επιπλέον δράσεις αλλά όπως είπε και ο κύριος Σταγιάν σήμερα το πρωί ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις γραμμές του προοδισμού που εμείς διαχειριζόμαστε για τα επόμενα τέσσερα έτη και για τις πολιετής προοπτικές θα πρέπει να εξετάσουμε και με άλλους συναδέλφους στην Επιτροπή το πώς θα μπορούσαμε να εδραιώσουμε όλες αυτές τις ε, ε, δημοσιονομικές δράσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ότο. Ο κύριος Σταγιάννη αναφέρθηκε σε αυτό που είχαμε πει για την ε, βιομηχανική κληρονομιά. Αν το περιλάβουμε δεν θα ήταν αντίθετος αυτό ισχύει ή διαφωνείτε. Ωραία. Ε, να πω ότι είναι σημαντικό να το ξέρει αυτό ο εισηγητής μας για τις γραμμές για τον τουρισμό. Αλλά νομίζω ότι αυτό αποτελεί και μια καλή λύση. Ντομινίκα, έχει το λόγο. Ωραία. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι Είδατε όλοι, είπατε περίπου όλοι τα ίδια. Δύο πράγματα μου προκάλεσαν εντύπωση. Ότι όλοι κάνουμε την ε, ίδια ανάλυση περίπου και δεύτερον ότι τέλος πάντων για τον προπολογισμό έχουμε τις ίδιες απόψεις. Να σας πω που βρισκόμαστε τώρα. Η Κομισιόν έκανε επιδρομή τέλος πάντων στα συρτάρια όπως λέμε και για το 2011 θα πρέπει να γίνει ακόμα δουλειά στον τομέα του τουρισμού. Το δεύτερο είναι ότι μου προκαλεί έκπληξη ο χαμηλός αριθμός βουλευτών γιατί είναι ανώφελο να δουλεύουμε εδώ στην Κομισιόν αν δεν βρίσκεται κάτι λειτουργικό που να μας υποστηρίζει η δουλειά μας αποβλέψτε να ανοίξουμε νέους δρόμους όσον αφορά τον έλεγχο, την ευθύνη και την ε, πρόθεση νέων πολιτικών. Αν αυτά οδηγήσουν τέλο πάντων σε ένα γκρεμό δημοσιονομικό, άσκοπη δουλειά. Και δεν το λέω αυτό επειδή κάνω την εισήγηση για τον προπολογισμό, αλλά θα πρέπει η Επιτροπή μας να συνειδητοποιεί ότι η πολιτική δουλειά θα είναι κενή αν δεν έχει τρόπους υλοποίησης. Τρίτο σχόλιο και τελευταίο τα περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα. Για το 2011 είδαμε ότι η Κομισιόν έκανε μια ισορροπιστική εργασία και αναζητούσε μέσα σε άλλες πολιτικές όπως την πολιτική των δικαιωμάτων των επιβατών, ασφάλεια που κάνουν οι υπηρεσίες κάνοντας ζητησία όμως στις δαπάνες των υπηρεσιών αυτών και η προσπάθεια αυτή φαίνεται ότι δεν αρκούσε για το TNT, αλλά το πάντων ήταν σημαντικό που έγινε. Τώρα βρισκόμαστε όμως στο τέλος ε, της δυνατότητα προσαρμογής για τις πολιτικές των μεταφορών. Αυτό που θα ήθελα να πω ήταν ότι πώς θα μπορούσαμε να πάμε παραπέρα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι το περιθώριο για το πλαφόν βρίσκεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ το οποίο δεν είναι τίποτα, γιατί σημαίνει δεν υπάρχει περιθώριο. Και είδατε ότι είχαμε και κριτική αυτές τις ε, προτάσεις, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Τώρα, το να κάνουμε μια αναζήτηση στα εργαλεία ευελιξίας, νομίζω ότι αυτό θα κάνει το καινοτόμο όσον αφορά αυτές τις πολιτικές, γιατί αυτά τα εργαλεία είναι πολύ περιορισμένα φέτος, εξάλλου στα πλαίσια του MFF θα έπρεπε να υπάρξει αναθεώρηση και δεν έγινε. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι εμεί τέλο πάντων ε, βρισκόμαστε πλάση στον τοίχο, έχουμε κάνει υπερβολή στα αστέρια, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλο περιθώριο. Οπότε, όπως είπαν σωστά και ειλικρινά από την Κομισιόν, είχαμε λιγότερα 20 ε, εκατομμύρια ευρώ λιγότερα για τι υπηρεσίε αυτέ του 2012. Ήδη δηλαδή έχουμε βάλει χέρι και στον προπολογισμό του 2012 για αυτέ τις υπηρεσίε. Όταν λοιπόν μιλάμε για υπηρεσίε, ή για γραφεία όπω τέλο πάντων ε, οδικέ μεταφορέ κτλ. τότε δεν ξέρουμε τι χρήματα θα υποστηρίξουμε ένα τέτοιο οργανισμό γιατί δεν υπάρχει ούτε σάλιο. Οπότε αυτό σημαίνει και βεβαίω συμμερίζουμε την άποψη του Προέδρου ότι εντάξει βεβαίω θα πρέπει να αυξήσουμε τις προσπαθίες μας, διαφορετικά εντάξει δεν ε, θα κάνουμε τίποτα. Όμως, αν δεν υπάρξουν νέες δυνατότητες όσον αφορά τους πόρους, επειδή ακριβώς δεν βρισκόμαστε στο πλαίσιο το γενικό του ε, προπολογισμού, θα κάνουμε από το 2012 και μετά. Και βεβαίως αυτό το θέμα θα συζητηθεί όλο και περισσότερο στην Επιτροπή του Υπολογισμού, αλλά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα πρέπει να βγούμε από την ορθοδοξία του πολιτικού πλαισίου και αν δεν υπάρχει ούτε η θέληση ούτε τα μέσα τότε δεν θα γίνει τίποτα και αυτό μπορεί να γίνει από φέτος γιατί ενδεχομένω δεν υπάρξει καν και αναθεώρηση του τους πλαισίου και υπενθυμίζω ο, το ταμείο που ανέφερε η Μαριέτα και ο Αντώνιο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επειδή θα υπάρξουν άλλα παρόμοια εργαλεία αντιμετωπίζει πρόβλημα σοβαρό τη στιγμή που λείπει μάλιστα και ένα ταμείο για τι μεταφορέ. Οπότε οι δράσει που θα αποφασίσουμε εδώ στην Επιτροπή θα εξαρτηθούν από αυτό, αλλά ακόμα και οι απλέ δράσει θα εξαρτηθούν από όλα αυτά. Βεβαίω η κατάσταση δεν είναι. Ε, δεν είμαστε σε απέλπιδα κατάσταση, αλλά η κατάσταση είναι σοβαρή και αυτό θα συζητηθεί νομίζω και στην Επιτροπή Μεταφορών. Θα πρέπει πάντως να κάνουμε κάτι πιο δραστήριο αν θέλουμε λοιπόν να παραμείνουμε στο τωρινό πλαίσιο και αν θέλουμε να υπάρξει τέλο πάντων απόφαση ή δέσμευση από το Συμβούλιο, τότε οι προοπτικέ είναι πολύ δύσκολε. Να πω και κάτι άλλο. Νομίζω στην Επιτροπή μα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι περιορισμοί που έχουμε αφορούν την καθημερινή μα δουλειά και ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να είμαστε στη θέση να δουλέψουμε. Διαφορετικά θα έχουμε κανένα χρηματοοικονομικό μέσο. Ευχαριστώ Ντομινίκ για αυτήν τη θαυμάσια εισήγηση. Δεν με ξαφνιάζει που λείπουν πολύ και πάλι η εμπειρία μου λέει ότι οι λίγοι μερακλείδες είναι που συζητάνε αυτά τα θέματα εδώ στην ομάδα αλλά αξιόλογα μάλλον και ενδιαφέρονταν αυτά τα θέματα και που αφορούν και την εισηγήσή σου. Είπες ότι έχουμε την παρουσίαση της νομοδότησης τον Ιούλιο, μετά συζήτηση στην Επιτροπή 2 του Σεπτέμβρη και μετά βέβαια έχουμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα και βεβαίως προσβλέπουμε στο σχέδιο της νομοδότησής σου μετά από όλα αυτά που ακούσαμε και σήμερα από του συμμετέχοντε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Επόμενο είμαι στην ημερήσια διάταξη. Η Επιτροπή που θέλει να σχολιάσει κάτι, ο κ. Μπονούτσι ή ο κ. Ότο, έχετε να πείτε τίποτα. Ο κ. Μπονούτσι. Ο κ. Μπονούτσι. Ένα σύντομο σχόλιο για να απαντήσω στην πρώτη παρέμβαση του κ. Λιμπεράτσκι. Η Κομισιόν σκέφτεται το πώς θα προωθήσει ένα καλύτερο συντονισμό με τη Γενική Διεύθυνση που διαχειρίζεται τα διευθυντικά ταμεία. Και είναι σε μόνιμο διάλογο παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να χρησιμοποιήσουμε την, το μοχλό των πιστώσεων. Αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αλλά είναι μια καθημερινή προσπάθεια. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στα διάφορα. Υπάρχει οσδήποτε βουλευτής που να έχει κάποιο θέμα να θέσει. Αν όχι, πέρα τη συνεδρίαση, υπενθυμίζω στους συντονιστές ότι έχουμε συνεδρίαση. Στους δύο συντονιστές που είναι παρόντες ότι θα συνεδριάσουμε στις 4.30. Αυτά ευχαριστώ. Πέρα συνεδρίαση.